ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε με τους αυξημένους πόρους να πετύχουμε τους στόχους ε, της ε, συνθήκης της Λισαβόνας και θέτει το θέμα της ελευθερίας των θεσμικών οργάνων μας όσον αφορά την πολιτική τους δράση με βάση τον προϋπολογισμό. Προτείνει απλούστευση των κοινών πολιτικών, την πολιτική συνοχής που έχει πολλά συνεισφέρει στο παρελθόν και θα συνεισφέρει στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει πρότυπο συνεννόησης και συνεργασίας λαών. Με το πολιετέ σε πλαίσιο ε, θα μπορέσουμε να περάσουμε σε μια νέα φάση πολιτική συνοχής μέσω των διάμεσων περιοχών. Προτείνουμε μια νέα αρχιτεκτονική του ε, Ταμείου που θα ενισχύσει την ισότητα ευκαιριών σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης άσχετα από την οικονομική κατάσταση ή τα μειονεκτήματά τους απέναντι στις πιο ανεπτυγμένες περιοχές άσχετα από τις ε, ευαισθησίες ή τα προβλήματα που έχουν σήμερα ή θα έχουν αύριο. Η συνοχή μεταξύ των διαφόρων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί βασικό στόχο. Στρατηγική κεντρική από τον οποίο εξαρτάται το ίδιο το μέλλον τη Ευρώπη. Οι προτάσει που υποβάλλονται είναι προ τη σωστή κατεύθυνση και αν γίνουν δεκτέ θα βοηθήσουν στο μέλλον. Κύριε Πρόεδρε, η ψηφοφορία στην έκθεση του κυρίου Γκαρίγκα θα αποτελέσει μια απλή επιλογή. Μια Ευρώπη που θα προχωρήσει, μια Ευρώπη αυτών που πέρα από τι πολιτικέ του πεπιθήσει είναι υπέρ του μέλλοντο τη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Η κυρία Ήλτα Φιγουρέιντο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι απαράδεκτο σε στιγμή τέτοια κρίση στη ζώνη ευρώ εξαιτία των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και τη έλλειψη αλληλεγγύη και οικονομική και κοινωνική συνοχή. Ε, είναι απαράδεκτο, λέω, ε, να μην συζητούμε για αλλαγή, ριζική αλλαγή των πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί όταν ζούμε μια τέτοια οικονομική κοινωνική και κοινωνική κρίση, χρειάζεται να αναζητήσουμε ένα καινούριο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο με σημαντική αύξηση του ευρωπαϊκού προπολογισμού για να υποστηριχθεί η οικονομική και κοινωνική συνοχή ε, με μείωση της ε, υποχρέωσης ε, ε, εθνικής συμμετοχή για τις ε, χώρες με τις πιο σημαντικές οικονομικές δυσκολίες έτσι ώστε αυτά τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν στην υποστήριξη της παραγωγής ε, στην ενίσχυση της απασχόλησης στην εκρίζωση της φτώχειας στη μείωση των κοινωνικών διαφορών και οποιονδήποτε διακρίσεων και ιδιαίτερος με βάση το φύλλο η υποστήριξη της ε, ανάπτυξης ε, και της ε, ειρήνης θα πρέπει επίσης να οδηγήσει σε μείωση των δαπανών άμυνας. Γι' αυτό το λόγο πιστεύουμε ότι η έκθεση αυτή δεν είναι αρκετή για να εξασφαλίσουμε ένα πιο δίκαιο μέλλον για την Ευρώπη και τους πολίτες της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Φιγκερέντο. Αντιλαμβάνεστε ότι ε, ε, αναλαμβάνοντας την Προεδρία της συνεδρίασης θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου για το θάνατο του Χόρχε Σεμπρούν ε, που έλαβε χώρα πριν από μερικές ε, ώρες στα 87 του απεβίωσε ήταν εχμάλωτος στο στρατόπεδο του Μπούχενβαλτ αντιμετώπισε τις γερμανικές δυνάμεις στην Γαλλία και το καθεστώς του Φράγκο στην Ισπανία ε, επίσης ε, ήταν ένας στρατευμένος, εξαιρετικός ε, στρατευμένος ε, συγγραφέας που είχε βραβευθεί με το βραβείο βιβλίο της χρονιάς του Ευρωκοινοβουλίου. Ήμουν φίλος του και σύντροφός του και θα ζητήσω από τον πρόεδρο Μπούζεκ να στείλει στους συγγενείς τους ένα μήνυμα συλληπιτήριο για το θάνατό του. por un για ένα λεπτό λόγο στον κύριο Φοντάνα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, βρισκόμαστε λοιπόν ε, σε μια πολύ κρίσιμη φάση της ιστορικής ε, τη οικονομική ιστορία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η επιτροπή, την οποία συστήσαμε κατά τη διάρκεια αυτού του έτου, αναμφίβολα διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο. Είμαστε κατά της αύξησης του προεπολισμού σε επίπεδο αρχής. Βέβαια πρέπει να δούμε πού μπορούν να γίνουν περικοπές. Γιατί πρέπει να γίνουν περικοπές στον ευρωπαϊκό προεπολισμό. Αυτή τη στιγμή τα ευρωπαϊκά κονδύλια δυστυχώς δεν χρησιμοποιούνται σωστά. Το αντίθετο συμβαίνει. Ίσως ε, στο θέμα της ε, χρήσης ε, των κονδυλίων πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες ε, να είναι τώρα πεπισμένοι για τη χρησιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς επιθυμούμε να στρέψουμε την προσοχή ε, σε πολλά κονδύλια ε, που διοχετεύονται στην πολιτική διεύθυνση. Πολλοί δεν ξέρουν που καταλήγουν αυτά ή για την ολοκλήρωση. Και αυτά δεν δίνουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και θέλουμε να επισημάνουμε το γεγονός ότι ορισμένες περιοχές μπορεί να είναι και εικονικές αυτές, δεν λαμβάνουν ποτέ τα κονδύλια. Και αν κάποιες άλλες περιοχές παίρνουν κάποια κονδύλια ή γίνεται κακή δική τους χρήση ή χρησιμοποιούν τα κονδύλια για όχι απόλυτα νόμιμους ε, τρόπους. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θέλουμε η Ευρώπη να ανακτήσει την αξιοπιστία της και μέσα από περικοπές. Ευχαριστώ πολύ. Ο, λίγος, ο λόγος του κύριο Φρανκ Βανέκη. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρώτο μου σχόλιο. Σε αυτή την έκθεση δεν βλέπω καθόλου προτάσεις για διαθωτικές περικοπές. Για παράδειγμα, ε, κατάργηση ε, περί των οργάνων όπως η Επιτροπή των Περιφερειών, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και μια σειρά άλλων ευρωπαϊκών γραφείων και υπηρεσιών. Δεν γίνεται καμία προσπάθεια να αναρωτηθούμε αν μήπως η Ευρώπη θα πρέπει ε, αν καταδικάζουμε την Ευρώπη ε, να ζει με ένα μεγάλο αριθμό ε, φόρων, για παράδειγμα. Αντιθέτως, θα έπρεπε οι φόροι να μειωθούν. Αν αυτή τη στιγμή γίνεται λόγος στην πραγματικότητα για αύξηση του φορολογικού βάρους στους Ευρωπαίους πολίτες. Και επίσης ε, αυτό που κάνουμε είναι ε, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ε, περιορίσουμε τα κράτη-μέλη στις αυξήσεις των δημοσιονομικών τους Ο κύριος Μαρινέσκου για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά έχει ανάγκη από μια σταθερή απάντηση εκ μέρους της Ευρώπης. Η στρατηγική του 2020 αποτελεί απάντηση ενίσχυσης της Ευρώπης. Η έκθεση που έχουμε ενώπιόν μας προσθέτει σε αυτή τη στρατηγική έναν κεντρικό ρόλο. Δεδομένου ότι η συνθήκη της Λισαβόνας έδωσε νέες αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά κράτη-μέλη χρειάστηκε να κάνουν δημοσιονομικές προσαρμογές και οι συνέπειες είναι βαριές για τους πληθυσμούς. Όμως χρειαζόμαστε μια αυξημένη προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη πρέπει η κοινή αγροτική πολιτική και η πολιτική συνοχής να διατηρηθούν σύμφωνα με την έκθεση τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με βάση το πι δελτα ε, Πρέπει επίσης ο προϋπολογισμός να χρησιμοποιηθεί με αποτελεσματικότητα και βεβαίως πρέπει να τηρηθούν τα κριτήρια της συνοχής και της συνεκτικότητας. Θα πρέπει η ανάπτυξη να εξασφαλίσει εξέλιξη όλων των άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών. Η νέα αυτή δομή, η επταετής περίοδος και η αυξημένη ευελιξία ε, θα επιτρέψουν στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό να προσαρμοστεί καλύτερα στις μελλοντικές αλλαγές. Το ίδιο ισχύει και για τους ίδιους πόρους που είναι απολύτως απαραίτητοι για να υποκατασταθούν οι εθνικές συνεισφορές. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε φιλόδοξου στόχου για την ανάπτυξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο αυτό Συμβούλιο θα πρέπει να μπορέσει να δεχτεί αύξηση κατά 5% γιατί αυτή είναι απολύτως απαραίτητη προπόθεση για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Το πι του μέλλοντο πρέπει να περάσει στην οικονομική ανάπτυξη και να φέρει την οικονομική σταθερότητα στην Ευρώπη. Στα συγχαρητήριά μου προς τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μαρινέσκου. Ο λόγος για τρία λεπτά στην κυρία Γκαρδιαθάβαλ Ρουβιάλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ε, επενώντας ε, το έργο του εισηγητή και των συναδέλφων της Επιτροπής ΣΟΥΡΕ. Ιδιαίτερα όμως θα ήθελα να επενέσω την ε, αποφασιστικότητα και την ε, επιθυμία να καταλήξουν σε μια ε, συνενετική έκθεση από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μια έκθεση όπως αυτή που παρουσιάζουμε σήμερα. Ε, είναι ο δικός χάρτης για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον αν θέλουμε να επιτύχουμε τους πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους που έχουμε θέσει τον εαυτό μας, αν θέλουμε να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις των επόμενων χρόνων είναι το σενάριό μας για να βγούμε από την κρίση. Και προκειμένου η στρατηγική μας για το μέλλον να είναι συνεπής ε, και να δώσει αποτελέσματα. Η Ευρώπη είναι περισσότερο από το σύνολο των 27 κρατών μελών. Ε, γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε αυτήν την έκθεση, αυτόν τον προπολογισμό. Τη χρειαζόμαστε επίσης για να πετύχουμε τους στόχους της χιλιετίας ε, και για να βοηθήσουμε τους γείτονές μας ε, στα νότια της Μεσογείου, στον αγώνα της για τη δημοκρατία. Τη χρειαζόμαστε αν θέλουμε να συνεχίσουμε να πολεμάμε στον, ε, στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης και ενοτομίας. Αν θέλουμε να επενδύσουμε στην εκπαίδευση, σε υποτροφίες εράσμους. Αν θέλουμε να έχουμε ένα εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης και αλληλεγγύης αν θέλουμε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε, υποστηρίζουμε τα διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών και ενέργεια. Με λίγα λόγια, αν, αν θέλουμε περισσότερη Ευρώπη, χρειαζόμαστε μεγαλύτερο προπολογισμό. Γι' αυτό το λόγο, στην έκθεση αυτή λέμε ότι χωρί τα επαρκή κονδύλια δεν μπορούμε να πετύχουμε του στόχου που έχουμε θέσει. Ξέρουμε ότι ορισμένα μέλη του Συμβουλίου δεν συμφωνούν με την αύξηση του προπολογισμού. Το ακούσαμε σήμερα. Ούτε ήταν υπέρ ακόμα και σε εποχέ οικονομικής ευμάρειας. Ακόμα και τότε ζητούσαν ε, περικοπές. Συνεπώς το Συμβούλιο, αν δεν θέλει, αν δεν συμφωνεί με αυτό προτείνουμε, ποιους στόχους θέλει να εγκαταλείψουμε. Όμω, λέμε και κάτι άλλο. Λέμε και πώς να χρηματοδοτήσουμε αυτές τις πολιτικές και θέτουμε το θέμα των ιδιών πόρων. Είναι μια συζήτηση η οποία θέλει να καταργήσει τα, ε, καταρρύψει τα επιχειρήματα των χωρών που λένε ότι είναι καθαροί συνεισφέροντε και να καταργήσει και τις επιστροφές. Υπάρχουν δύο εναλλακτικέ λύσει βέβαια. Ε, την, αυτή που υποστηρίζω εγώ είναι ο φόρο των χρηματοοικονομικών συναλλαγών ο φόρος Ρομπέν των δασών, όπως ε, λένε ορισμένοι, που θα εξασφαλίσει 300 δισεκατομμύρια ευρώ στον προπολογισμό, ε, θα τιμωρήσει τους κερδοσκόπους ε, και θα αποφύγει να παίζονται παιχνίδια εις βάρον μας. Ένας τέτοιος φόρος θα εξασφαλίζε διαφάνεια και δεν θα επηρέαζε τους πολίτες μας, διότι θα ανάγκαζε να πληρώσουν αυτοί που δημιούργησαν την κρίση. Ένα πράγμα θέλω να πω, μεγαλύτερη φιλοδοξία για να πετύχουμε το ευρωπαϊκό σχέδιο να συνεχίσει το δρόμο του και να μην μείνει στάσιμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Έντερ. Ο λόγος για ένα λεπτό στον κύριο Αλεξάνδρα Άλβαρο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, εγώ γεννήθηκα το 1975. Τότε είχαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση καθόρισε τη ζωή μου. Ε, σήμερα με πονάει πάρα πολύ το ότι αναγκαζόμαστε να βάλουμε νερό στο κρασί μας. Όταν μιλάμε για αυξήσεις, ε, κατ' ουσίαν, τι σημαίνει αυτό, ότι δεν θέλουμε να κάνουμε μια ουσιαστική συζήτηση για τους ίδιους πόρους. Εγώ την έκθεση που είναι μια φιλόδοξη έκθεση και επιθυμεί να συγκεντρώσει την πλειοψηφία των ευρωλεπτών, εγώ δεν τη θεωρώ φιλόδοξη, ε, δεν σε ε, ε, το γεωργικό και το Ταμείο και το Ταμείο Διαρθρωτικών Αλλαγών. Ε, το μόνο που ε, αναφέρεται είναι τα χρήματα και λένε λείπουν χρήματα. Αλλά δεν αναφέρεται πού θα βρούμε τα περισσότερα κονδύλια. Δεν αναφέρονται καν οι διπόροι, ούτε και ορίζονται οι διπόροι. Αν πραγματικά θέλαμε διαρθρωτικέ αλλαγέ, τότε θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε την πρόταση του κυρίου Κάμερον, να κάνουμε ένα βήμα προ τα μπρο και να πούμε παγώνουμε του ίδιου πόρου, όμω Συμβούλιο ζητάμε οι μη χρησιμοποιηθέντε ήδη πόροι να μπορούν να μεταφέρονται στην επόμενη χρονιά έτσι ώστε να χρηματοδοτούνται προγράμματα του μέλλοντος και να γίνονται περικοπές. Κυρίες και κύριοι, ε, δεν μπορούμε να μετρήσουμε το μέλλον της Ευρώπης ε, με δεκαδικούς αριθμούς και για το λόγο αυτό εγώ πρέπει να σας πω ότι είμαι απογοητευμένος όσον αφορά στην έκθεση που έχει κατατεθεί. Και σήμερα το πρωί ο κύριος Δόλ ήρθε σε τρέχοντας να μιλήσει στην Ολομέλεια για την ανάγκη αυξημένου προϋπολογισμού, αλλά έτρεξε τόσο γρήγορα που λαχάνιασε και δεν μπορούσε να μιλήσει. Ακριβώς αυτό δείχνει τη συζήτηση για τον πολιετή προϋπολογισμό. Ο Ευρωπαϊκό Προπολογισμό είναι το 1% περίπου του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο ότι θέλουμε πιο πολλά λεφτά, δεν φτάνει. Όμω η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να δαπανίσει τα διαθέσιμα χρήματα εκατομμύρια επί εκατομμυρίων στα ε, περιφερειακά ταμεία και Ταμείου Ταμείο μένουν να χρησιμοποιείται και επιστρέφονται στα... Ε, και άρα γιατί χρειάζεστε περισσότερα λεφτά αν δεν μπορείτε να ξοδέψετε ούτε αυτά που έχετε. Εδώ σε αυτό το Κοινοβούλιο έχουμε κάποια προβλήματα. Ο ε, οι αρχηγοί, ο κύριος Ντόλ, ο κύριος ε, Σούλτς και άλλοι έφυγαν, δεν είναι εδώ, για να μιλήσουν περισσότερο για την ποιότητα και όχι για την ποσότητα. Ας πούμε, η, τα Ταμείο Συνοχής για τις πιο φτωχές περιοχές που πρέπει να πάει το 30% την καινοτομία και σε άλλους χώρους. Αλλά οι παυλόφ της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ε, θα πέσουν πάνω στον, στο τείχος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αυτής της χρονιάς. Παρακαλώ να σέβεστε τον, το χρόνο. Ε, Τώρα βέβαια είναι η σειρά τη κύρια Ντουράν και λυπάμαι που το λέω αυτό, αλλά αν δεν σεβόμαστε το χρόνο μα δεν θα καταφέρουμε να τελειώσουμε έγκαιρα. Ο λόγο στην κυρία Ντουράν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για λόγους και ταυτόσιμους αλλά και διαφορετικούς αλλά λόγους που έχουν επιβαρυνθεί από την κρίση οι, εθνικοί προϋπολογισμοί προφανώς ε, έχουν δυσκολίες όποιες και αν είναι οι κυβερνήσεις γίνονται προσπάθειες σε δημοσιονομικό επίπεδο και έχουμε δύο εναλλακτικέ. πρώτον να φέρουμε μόνοι μας τις απαραίτητες προσπάθειες με διαφορετικούς βαθμούς επιτυχίας περικόπτοντας ή έσοδα, αυξάνοντας έσοδα ή περικόπτοντας δαπάνες και ε, ε, κάνουμε ε, μια κατάσταση περιοκόπτοντας Η εσοδα αυξανοντας εσοδα η τα δαπανες εναλλακτική είναι αυτή που θα στηρίξω. Είναι η συγκέντρωση και η, των πόρων και η αλληλεγγύη. Να παίξουμε μαζί το, στην, σε πεδίο δημοσιονομικής αλληλεγγύης και ε, για να επιβληθεί ένας φόρος ε, ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Υπάρχει αυτή η περίφημη σύμβαση που επιβάλαμε στη διάρκεια της, υποβάλαμε στη διάρκεια της διαβούλευσης στο Συμβούλιο και εδώ θα πρέπει όλοι μαζί, κυβερνήσεις, κοινοβούλια κλπ. να συγκεντρώσουμε τις προσπάθειές μας για να δουλήσουμε ε, να δουλέψουμε με αλληλεγγύη. Δεν μπορούμε να έχουμε και το σκύλο χορτάτο και την πίτα γερή. Δεν μπορούμε να προσφέρουμε λιγότερα και να παίρνουμε περισσότερα. Άρα θεωρώ ότι αυτή η σύμβαση, το σύστημα διαλόγου μεταξύ κυβερνήσεων Ευρωπαϊκή Ένωση, Εθνικά Κοινοβούλια και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ο καλύτερο τρόπο για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό έργο, στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Ευχαριστώ, Ιζαμπέλ. Για ένα λεπτό, λόγο στον κύριο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή είναι κάκιστη. Θα μπορούσαμε να την ε, πετάξουμε κατευθείαν στα σκουπίδια. Οι πολίτες μας αντιμετωπίζουν οδυνηρότατα ε, μέτρα λιτότητας και είναι παράλογο εμείς να ζητούμε μεγαλύτερο προπολογισμό να δαπανηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι δυνατόν να απορροφούμε κονδύλια αριστερά-δεξιά πρέπει να εστιαστούμε στα φτωχα κρατημέλη, θα πρέπει να εξετάσουμε project καινοτόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά τα κρατη για να τα βοηθήσουμε. Εμείς λέμε όμως με αυτή την έκθεση ότι χρειάζονται περισσότερα χρήματα στα διορθωτικά προγράμματα, στα διορθωτικά ταμεία. Πάντα η ίδια παλιά ιστορία. Δεν μιλούμε για την αποτελεσματικότητα, για τη σωστή διαχείριση και τη σωστή δαπάνη των ποσών. Αυτή τη στιγμή αφήνουμε παράλληλους ανθρώπους, ανθρώπους με αναπηρίες στο κρύο. Ε, όχι, χρειαζόμαστε καλύτερη δαπάνη των ποσών. Ένα λεπτό για τον κύριο Μοργάντη. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να υπογραμμίσω ορισμένα στοιχεία αυτή τη τόσο σημαντική έκθεση, ξεκινώντα από το σύστημα εισόδων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι απόλυτα σαφέ ότι ο μηχανισμό που ισχύει τώρα ε, είναι ασυνεπή ε, με πάρα πολλά θέματα αρχή, όπω οι βρετανικέ επιστροφέ. Εξάλλου, ο μηχανισμό εισόδων τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι καθόλου διαφανή. Στο σημείο αυτό, νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να έχουμε ένα σύστημα ιδίων πόρων, ή θα ήταν καλύτερα να έχουμε ένα ενοποιημένο σύστημα, ε, παραδείγματο χάρη για το ΦΠΑ. Είναι σαφέ ότι οι Ευρωπαίοι πολίτε δεν θα πρέπει να πληγούν από περαιτέρω βάρη. Η Ευρώπη ε, μπορεί να αντικαταστήσει τα κράτη-μέλη σε θέματα φορολογικά. Ε, στην έκθεση αναφέρονται διάφορε προτεραιότητε, ορισμένε εξ αυτών είναι σημαντικέ, αλλά παρόλα αυτά όλε είναι ιδιαίτερα δαπανηρέ. Αναφέρονται τα project bond και τα ευρωομόλογα. Ε, όσον αφορά αυτά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να μην δημιουργήσουμε περαιτέρω χρέο. Εμεί ω Ευρωπαίοι, ε, ω Ευρωβουλευτέ ε, μπορούμε να βελτιώσουμε το θέμα των εσόδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξοικονομήσουμε πολλά εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και αυτό δεν είναι απλά λόγια, δεν είναι λαϊκίστικες κουβέντες. Τον διάκοψε δυστυχώς ο πρόεδρος, τον ομιλητή. Ο λόγος στην κυρία Ντότζη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Επίτροπε ο κύριος Φερχόφστατ μας εξήγησε γιατί η Βρετανία πρέπει να δώσει περισσότερα χρήματα και περισσότερες εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μας δείχνει ακόμα μια φορά το τρόπο με τον οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο, η εθνική του κυβέρνηση και οι πολίτες ε, αντιμετωπίζονται από μερικού. Αυτό που δεν είπε ο κύριος Φερχόφστατ γιατί φοβήθηκε είναι ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο οι επιχειρήσεις είναι αναγκασμένες να δαπανίσουν 30 εκατομμύρια λίρες για να συνάδουν με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους και θα, ενώ οι ψαράδες θα θέλανε τα 3,3 να τα έχουν στην τσέπη τους αυτά που έχουν χάσει όταν η Ευρωπαϊκή τα, οι ψαράδες από την Ευρωπαϊκή Ένωση έρχονται στα χωρικά τους ύδατα. Δεν αποτελεί επανάληψη εθνικού προπολογισμού, κοινοτικό προπολογισμό μας λέτε. Όμως δεν μπορείτε να τον διαχωρίσετε από την πραγματικότητα των πολιτών. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία συνεισφορά 6,4 δις και θα ξεπεράσει τα 10 αν δεν υπάρχει αυτή η επιστροφή. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο αυξάνοντας του φόρου, περιορίζοντα τι υπηρεσίε ε, για τα σχολεία κλπ. Δεν έχετε άλλο χρόνο. Το λόγο έχει ο κύριο Κάρα για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ε, πέντε ερωτήματα πρέπει να υποβάλουμε τι είδου προπλογισμό χρειάζεται η στρατηγική ανάπτυξη και απασχόληση του 2020. Δεύτερον, τι είδου προπολογισμό χρειάζεται η νομισματική ένωση. Τρίτον, τι είδου δυνατότητε εξοικονόμηση υπάρχουν. Τέταρτον, τι είδου προπολογισμό χρειάζονται τα ενωμένα κράτη τη Ευρώπη. Πέμπτον, ποιο είναι ο ρόλο που μπορεί και πρέπει να παίξει η Ευρώπη το 2020. Μα και θέλουμε να παίξουμε ρόλο μέχρι το 2020. Εμεί, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναλαμβάνουμε με τις ευθύνες μας, ε, λέμε τα πράγματα με το όνομά της. Ε, στην Αυστρία θα έλεγα ε, χωρίς λεφτά δεν χορεύει το αρκούδι. Εμείς λοιπόν ε, ε, θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις ε, προκλήσεις. Επιθυμούμε να είμαστε περισσότερο ανταγωνιστικοί, να έχουμε περισσότερο βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση, έρευνα, ολοκλήρωση. Μα όλα αυτά δεν μπορούν να υλοποιηθούν με λιγότερα χρήματα, χωρίς αξιολόγηση των κονδυλίων, χωρίς να υπάρχει το σύστημα των ιδιών πόρων. Η περισσότερη Ευρώπη δημιουργεί και ένα δυναμικό σημαντικό Εξοικονόμηση κονδυλίων στα κράτη-μέλη. Η περισσότερη Ευρώπη ε, δημιουργεί, είναι πιο αποτελεσματική και είναι η δική μας η απάντηση στην παγκοσμιοποίηση, στο μέλλον, ε, στα δημόσια χρέη. Μα τι θέλουμε επιτέλους θέλουμε να μην παγώσουμε τον προεπλογισμό. Όποιος παγώσει τον προεπλογισμό θα ζημιώσει την Ευρώπη και θα αποδυναμώσει εμάς στις προσπάθειές μας για την υλοποίηση των ονείρων των Ευρωπαίων πολιτών. Ε, πολλοί ε, θέλουν να αντιμετωπίσουν ε, τον φόρο χρηματοψηφιτικών συναλλαγών στο πλαίσιο των ιδίων πόρων. Ας το αντιμετωπίσουμε αυτό σοβαρά και να μην στρουθοκαμιλίζουμε ας ε, αναλάβουμε τις ευθύνες μας και ας ε, εγκρίνουμε την έκθεση, ας την υπερψηφίσουμε. Για τρία λεπτά ο λόγος στον κύριο Κάλφιν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η έκθεση Γκαρίγα κάνει λόγο πιο πολύ για πολιτική παρά για οικονομία. Και ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Χάου και όλου του άλλου συναδέλφου που πραγματικά εστίασαν την έκθεση στην πολιτική. Ε, τα κονδύλια είναι μέσον για την επίτευξη στόχων. Οι πολιτικές είναι αυτές που μετράνε και πρέπει να συζητηθούν στο πλαίσιο του νέου ΔΕΛΤΑΠ. όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης περνούν από μια εποχή λιτότητα και παίρνουν μέτρα λιτότητας. Αυτά τα μέτρα σχετίζονται επίση με την καταπολέμηση τη κρίσης. Και αυτή την κρίση μπορούμε να την πολεμήσουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με τη ρύθμιση των χρηματοοικονομικών αγορών, με τα αναπτυξιακά προγράμματα. Όλα αυτά είναι μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που μπορούν να βοηθήσουν αυτά που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο. Συνεπώς δεν υπάρχει κάποια αντίφαση μεταξύ αυτών των δύο, ούτε κάποια σύγκρουση. Η ενίσχυση της Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ε, προστιθέμενη αξία. Αυτή η προστιθέμενη αξία και η αλληλεγγύη δεν είναι κενές λέξεις. Πρέπει να εξηγήσουμε στους φορολογούμενους ότι δεν τους ζητάμε απλώς να πληρώσουν περισσότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι η Πολωνία και η Βουλγαρία βρίσκονται στην ίδια αγορά, αλλά είναι πιο φτωχέ χώρε. Πρέπει να ανταγωνιστούν πιο πλούσιου εταίρου και πρέπει να του βοηθήσουμε. Η αλληλεγγύη έχει πολλά πρόσωπα και αυτά έχουν σχέση με, την προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής, με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια. Δεν μπορούμε να ε, επιτύχουμε στην, στον τομέα της επιστήμης, στον τομέα της έρευνας, στον τομέα της ενέργειας, χωρίς κοινέ ευρωπαϊκές πολιτικές. Και ασφαλώς υπάρχουν συγκυρίες, συγκεκριμένε συγκυρίες, οι οποίες είναι ρευστέ. Θα πρέπει να τι ε, λάβουμε υπόψη. Αλλά αποτελέσματα. Αλλά δεν είναι δυνατόν στην πολιτική συνοχή να βάλουμε όλα τα άλλα, όλες τις άλλε ανάγκε των άλλων πολιτικών, ε, ενέργεια, ε, δικτύων κλπ η μείωση των κονδυλίων για υπάρχοντα, από υπάρχοντα κονδύλια, από υπάρχοντα προγράμματα δεν θα βοηθήσει. Δεν θα καταφέρουμε έτσι να δώσουμε προστιθέμενη αξία στους ε, φορολογούμενους μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια κοινοτική μέθοδο, έχει ένα σύστημα για το νόμισμα, για τις αγορές αυτό το 5% δεν αρκεί καν για να λύσουμε όλα μας τα προβλήματα. Θα πρέπει να δούμε και τα Eurobond και, τα, ε, και τις άλλες εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης. Ευχαριστώ πολύ. Ένα, ένα λεπτό για την κυρία Πάουλσεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τελικά κατέληξε ο συμπέρασμα ότι η δουλειά της Σούρα ήταν ό,τι καλύτερο είδα ποτέ. Γιατί ό,τι είναι καλό για το μέλλον της Ευρώπης περιλαμβάνεται σε αυτή την έκθεση της Επιτροπής Σούρε. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πω ότι εγώ προσωπικά ανησυχώ τα μάλα για αυτά που δεν πράξαμε. Και τι δεν πράξαμε να ορίσουμε προτεραιότητες Βεβαίως και αναφερόμαστε σε όλες τις νέες προκλήσεις, όμως δυστυχώς ε, διατηρούμε και τις αγκυλώσεις ε, του παρελθόντος. Και βεβαίως δεν μπορεί να έχει κανείς και το σκύλο και την πίτα και το σκυλοχορτάτο και την πίτα ολόκληρη. Θα έπρεπε λοιπόν να είμαστε πολύ σκληρότεροι από ό,τι αποδειχθήκαμε. Και εκείνο που με ανησυχεί περισσότερο είναι το γεγονός ότι τις προτεραιότητες αυτές τις αφήσαμε να τις ορίσει το Συμβούλιο. Αυτό λοιπόν δεν είναι καλή κληρονομιά για το μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Κάλαναν. Κύριε Πρόεδρε οι φορολογούμενοι στην Ευρώπη που κερδίζουν τα χρήματά τους με τέτοια δυσκολία επιθυμούν η Ευρώπη να κάνει λιγότερα και να κάνει περισσότερα. Επιθυμούν να στηρίξουν το ευρωπαϊκό προπλογισμό, ο οποίος είτε μας αρέσει είτε όχι θα λαμβάνει υπόψη του ότι ζούμε σε εποχή λιτότητας. Θέλουν η Ευρώπη να εστιάζει την προσοχή της σε λίγους τομείς όπου πραγματικά η Ευρώπη μπορεί να προσθέσει υπεραξία και τις υπόλοιπες δραστηριότητες να τις αφήσει στα κράτη-μέλη. Δυστυχώς η έκθεση αυτή δεν προτείνει τίποτα από όλα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είναι σαφές πρόταση αυτή αύξηση του 5% είναι απαράδεκτη. Η ιδέα των περίφημων ιδίων πόρων, μα και αυτή παντελώ απαράδεκτη, ε, απλά είναι ένα τέχνασμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο προπολογισμό πρέπει να εξυγχρονιστεί, να υπάρξει ανακατανομή κονδυλίων για να έχουμε μέλη, ε, ωφέλη στο μέλλον ε, και όχι ζημιέ όπω το παρελθόν. Ε, οι χώρε που ήθελαν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά είχαν προβλήματα και αναγκάστηκαν προσπαθήκαμε να τις διασώσουμε, λάθος ήταν αυτό. Στο μέλλον λοιπόν ε, βλέπουμε ότι δυστυχώς δεν θα γίνουν πολλά πράγματα και γι' αυτό την έκθεση αυτή πρέπει να την απορρίψουμε. Ευχαριστούμε κύριε Κάλαμαν. Το λόγο έχει ο κύριος Λάσλο Σούριαν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ίσως η πλέον βασική έκθεση είναι αυτή που μας απασχολεί τώρα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το πρώτο το οποίο εκφράζει τις σκέψεις ε, μας για τα επόμενα 7 χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να προβάλλει προτάσεις, γιατί αυτό είναι ο μόνος τρόπος για να φτιάσουμε σε συμφωνία και να αποφύγουμε σκάνδαλα τύπου απόρριψης των προσχεδίων του Συμβουλίου. Σημασία έχει να ξέρουμε τι αποζητούμε και μπορούμε όλα αυτά να τα εντάξουμε στον τρόπο σκέψης των άλλων. Υπάρχουν ορισμένα σημεία που θα μας απασχολήσουν στην συνθήκη της Λισαβόνας πριν εκφραστούν σοβαρές επικρίσεις. Θα πρέπει να δούμε πώς θα ορίσουμε το θέμα των ιδίων πόρων. Θα πρέπει να περάσει και αυτό το μήνυμα ότι δηλαδή μία μικρή αύξηση χρειάζεται στον προϋπολογισμό γιατί θα πρέπει να μας απασχολήσει και ο πληθωρισμός και να δούμε πώς θα επιδράσει στο όλο δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν μιλάμε για μεγάλο ρυθμό ανάπτυξης. Μιλάμε για σοβαρές δαπάνες δυνάμει των διαρθρωτικών ταμείων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να περικοπούν τα κονδύλια των ταμείων. Ο Μίκλος Ζίνερη το 1600 η Ουγγρικής και Κροατικής καταγωγής είχε πει ε, μην πλήξετε τον Ούγγρο, θοπεύσετε τον. Το ίδιο μπορώ να πω για την ΚΑΠ, διότι αν πλήξετε την ΚΑΠ δεν σημαίνει ότι πλήττετε μόνο τους Ρουμάνους, τους Ούγγρους και ούτω καθεξής, αλλά πλήττετε όλες τις χώρες της Ευρώπης γιατί όταν είναι ε, η εκλογική βάση συγκεκριμένη πάντα πλήττουμε και τους πολίτες μας. Έχουμε μεγάλες πολιτικές ομάδες πίσω μας και θα πρέπει να εκπροσωπήσουμε τους πολίτες μας. Έλεξε ο χρόνος σας. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή και τον Πρόεδρο για τη δουλειά που έχουν κάνει επί της έκθεσης αυτής. Η συζήτηση σημερινή τονίζει πως θα γίνει μάχη στο Συμβούλιο ε, για πολλά θέματα, μεταξύ των οποίων τη συνολική αύξηση, τη Βρετανική επιστροφή και τους ίδιους πόρους. Και για να είμαστε δίκαιοι, πέρα από το ζήτημα της ε, Βρετανικής επιστροφής, όπου θα είναι μόνοι τους οι Βρετανοί. Νομίζω πως το Κοινοβούλιο προσπάθησε να επιτύχει κάποιους συμβασμούς και βεβαίως όταν μιλάμε για τόσο πολύπλοκες εκθέσεις αυτό είναι αναπόφευκτο αλλά κάποιους από τους συμβασμούς τους καλωσορίζω για την διάρκεια ας πούμε και την δομή των επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών. Επίσης τον συμβιβασμό για την πολιτική συνοχής Πιστεύω πως η πολιτική συνοχή έχει ζωτική σημασία αν είναι να έχουμε δουλειές και ανάπτυξη στην Ένωση πέρα από το 2013. Οπότε χρειάζεται επαρκής χρηματοδότηση τουλάχιστον στο επίπεδο το τωρινό αν όχι και περισσότερο στο μέλλον. Οι επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές πρέπει να αφορούν τι δουλειές και την ανάπτυξη εάν είναι να αφορούν τους πολίτες. Οπότε, πέρα από την πολιτική συνοχή, πρέπει να χρηματοδοτήσουμε την έρευνα και την ανάπτυξη στα πανεπιστήμια και τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. οπότε πρέπει να χρηματοδοτήσουμε παρκώ το πρόγραμμα πλαίσιο 8. Η υποδομή τη Ευρωπαϊκή Ένωση επίση αποτελεί αντικείμενο επένδυση. Μεταφορέ, ενέργεια, ευρυζωνικότητα σε περιοχέ τη υπαίθρου και βεβαίω και οι περιοχέ τη υπαίθρου δεν πρέπει να τι ε, ξεχάσουμε. Για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται κάποιος μηχανισμός και εταίροι για ένα λεπτό έχει το λόγο η κυρία Ρίκα Μάνερ. Ευχαριστώ πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν να συγχαρώ τον εισηγητή για την εξαιρετική αυτή έκθεση και την εξαιρετική του εργασία στην Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή. Όταν μιλάμε για το δημοσιονομικό αυτό πλαίσιο, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να έχουμε τα κατάλληλα μέσα για να επιτύχουμε τους στόχους της στρατηγικής 2020. Σε αυτή την έκθεση ορίζεται ότι αν δεν υπάρχει ένας δυνατός προϋπολογισμός και μεγάλη συνοχή στην ΚΑΠ, δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτούς τους στόχους, διότι αυτό είναι το μόνο μέσο που διαθέτουμε για να δημιουργήσουμε εργασία και ανάπτυξη. Θα πρέπει να περάσουμε αυτά τα σαφή μηνύματα και θα πρέπει να αναπτυχθούν και σε άλλους τομείς. Κύριε Επίτροπε, θα πρέπει να λάβετε υπόψη αυτές τις απαιτήσει που προβάλλει το Κοινοβούλιο ως προς το δημοσιονομικό πλαίσιο και την ΚΑΠ. Στην έκθεση επίσης λέμε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη περιοχές, ιδιαίτερες περιοχές που πλήττονται ιδιαίτερα στον Βορρά. Έχει το λόγο για ένα λεπτό ο κύριος Βαντάλεν. Κύριε Πρόεδρε, η λέξη κλειδί για την Ευρώπη είναι εμπιστοσύνη. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και ειδικά το Κοινοβούλιο πρέπει να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών. Πώ θα γίνει αυτό, Πρώτον, όχι περισσότερη Ευρώπη ή περισσότερα λεφτά για την Ευρώπη, αλλά καλύτερη Ευρώπη. Ευρώπη με προσθέμενη αξία και να μην ασχολούνται η Ευρώπη με πράγματα που μια χαρά μπορούν να κάνουν τα κρατημέλη όπως ο αθλητισμός ή ο τουρισμός. Δεύτερον, το Ταμείο Συνοχής να χρησιμοποιηθεί για τις πραγματικά φτωχές περιοχές της Ευρώπης. 50% πάει αυτή τη στιγμή σε πλούσια κρατημέλη όπως η Γαλλία και η Γερμανία. Απαράδεκτο. Και αν τα ρυθμίσουμε σωστά δεν θα χρειάζεται να κάνουν τα λεφτά κύκλους άσκοπους. Τρίτον, να επενδύσουμε στην γεωργία και την βιομηχανία του μέλλοντος. Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση υπολέδω είναι αποτυχία. Πρέπει να πληρώνει ο πολίτης χωρίς να επωφελείται καθόλου. Εντάξει, καλή σας όρεξη, αλλά προσοχή στην κατάσταση. Ο κύριος Φερνάντες έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την εξαιρετική του έκθεση, διότι μας επιτρέπει μια καλή αρχή στην οικοδόμηση του νέου δημοσιονομικού πολιετούς πλαισίου, κάτι το οποίο θα συνδράμει το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Πρόκειται για μια φιλόδοξη έκθεση, αλλά και ρεαλιστική παράλληλα. Νομίζω ότι όλα τα θεσμικά όργανα έμαθαν το, πήραν το μάθημα από τη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση. Είμαστε μια ενωμένη Ευρώπη, αλληλέγγυα Ευρώπη και προσπαθούμε να συγκλίνουμε τις πολιτικές μας. Ελπίζω λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τις ε, μεγάλες προκλήσεις του μέλλοντος. Θα πρέπει να υπάρχει υπεροχή του κοινοτικού χαρακτήρα υπολογισμού και να ενισχύσουμε τον προϋπολογισμό. Η στρατηγική του 2020 είναι μια συνενετική στρατηγική. Θα πρέπει η στόχη αυτή να είναι μετρήσιμη μέσα στα πλαίσια των δημοσιονομικών πρόπτικων. Αυτή όμως η στρατηγική θα επιτύχει εάν λάβουμε υπόψη αυτές τις ε, δράσεις με βάση τους απότερους στόχους. Άρα το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να λάβει υπόψη την ε, μελλοντική στρατηγική 2020. Επίσης, βασιζόμαστε στην αρχή της αλληλεγγύης. Θα πρέπει η συνοχή να είναι οικονομική, περιφερειακή και εδαφική, καθώς και κοινωνική, έτσι ώστε να διαθέτουμε τα κατάλληλα κονδύλια για να καλύψουμε και την ΚΑΠ μεταξύ άλλων. Θα πρέπει να προωθήσουμε ένα πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο όπου τα έσοδα να μην εξαρτώνται κατά 80% από τους εθνικούς πόρους. Ευχαριστούμε. Η κυρία Κίνγκα Γκένς έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κρίση μας υποχρεώνει να αναθεωρήσουμε τις ιδέες μας για τους εθνικούς αλλά και για τον κοινοτικό προϋπολογισμό για να διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει των αναπτυξιακών στόχων και πρέπει επίσης να δούμε κατά πόσον η αναθεώρηση αυτή προσθέτει κάτι στα κεκτημένα. Είναι κάτι που δεν το έχουμε ακόμη πει και που αφορά τη συμβολή της συνθήκης της Λισαβόνας στο θέμα της εθνικής δικαιοδοσίας ως προς τη δικαστική συνεργασία. Θα θέλαμε εδώ και εδώ να σημειωθούν πρόοδοι. Πρέπει να επιτευχθεί επαρκής χρηματοδότηση του προγράμματος της Στοκχόλμης έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις μεταναστευτικές ροές και γι' αυτό χρειάζονται πόροι, πρόσθετοι πόροι. Τα τελευταία γεγονότα στη Βόρεια Αφρική μας υποχρεώνουν επίσης να αναθεωρήσουμε τη μεταναστευτική μας πολιτική. Και αυτό δείχνει ότι χρειάζεται μια συμπερίληψη και ολοκλήρωση και στη χρηματοδότηση καθώς και επίδειξη μεγαλύτερης ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, περισσότερης ευρωπαϊκής αλληλεγγύης για να μπορέσουμε να προασπίσουμε τις αξίες μας, να καταπολεμήσουμε την άνηση μεταχείριση και γι' αυτό χρειάζονται πόροι. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει η απλοποίηση του τρόπου κατανομής και χρήσης των πόρων αυτών που αυτή τη στιγμή γίνονται με ένα πολύπλοκο σύστημα και να υπάρχουν όλοι οι ίδιοι πόροι που χρειαζόμαστε για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί για την Ευρώπη. Ευχαριστούμε Κίνγκα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω το σχετικό άρθρο του κανονισμού που λέει, που αναφέρει ότι από τα θεωρία θα πρέπει όλοι οι παρατηρητές να παραμείνουν ήσυχοι και να παρακολουθούν τα δρόμενα. Θα ήθελα λοιπόν να μην υπάρχουν αντιδράσεις Άρα θα πρέπει παρακαλώ το προσωπικό να επιβλέψει ποιος χειροκροτεί και ποιος όχι, ποιος αντιδρά γενικότερα, διότι αυτό απαγορεύεται. Γι' αυτό να γνωρίζουν οι παρατηρητές τα θεωρία ότι όποιος αντιδρά θα πρέπει να απομακρυνθεί από την αίθουσα. Ο κύριος Έλλης έχει το λόγο. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στον εισηγητή για τη δουλειά που έχει κάνει τρομερή όσον αφορά το να επιτύχει συνένεση τρεις τομείς στους οποίους θα ήθελα να υποστηρίξετε τροπολογίες. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε πενταετής ε, οικονομικές προοπτικές. Αν μιλάμε για το 2020 θα πρέπει οπωσδήποτε οι επόμενες να είναι για πέντε χρόνια. Δεύτερον, δεν έχουμε δει τι γίνεται με την διαβεβαίωση του ελεγκτικού συνεδρίου. Όσοι ζητάνε περισσότερα λεφτά θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό ευκολότερα εάν ξέραμε απολύτως πού πηγαίνουν τα λεφτά. Και τέλος, για να απαντήσω στον κύριο Φερχόφστατ, δεν είναι σωστό να ξεχωρίζουμε ένα κράτο μέλο όταν είναι πολλά τα κρατημέλη που είναι καθαροί εισφορεί στον προπολογισμό. Εγώ θα έλεγα πω θα έπρεπε να υπάρχει ένα όριο ως ποσοστό του ΑΕΠ στην εισφορά στον προπολογισμό. Γιατί δεν είναι δυνατόν να διπλασιάζει τη εισφορά κρατών μελών σε καιρού λιτότητα. Ο κύριος Πίπερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. η αύξηση κατά 5% είναι δικαιολογημένη. Υπάρχει εξωτερική υπηρεσία, καταπολέμηση τρομοκρατίας, επένδυση στι υποδομέ και τελικά είναι δικαιολογημένη αυτή η απέτηση του Κοινοβουλίου. όμω το Κοινοβούλιο με την έκθεση Καρίγα χάνει και μια ευκαιρία γιατί θα ήμασταν ακόμη πιο αξιόπιστοι αν μπορούσαμε να δείξουμε πού μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική η Ευρώπη, πού μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα. Βλέπετε πως έχουμε πάρα πολλές ε, εξωτερικές ε, υπηρεσίες που κοστίζουν πάρα πολύ. Επίσης στη Γεωργία όπου κάποια κράτη-μέλη ακόμα δεν έχουν ε, καταφέρει να φτάσουν πιο κοντά στις συνθήκες αγοράς. Επίσης για την διαρθρωτική πολιτική θα συμπεριλάβω και την πολιτική συνοχή. Ευτυχώ πάρα πολλέ περιοχέ κατάφεραν να ξεπεράσουν το κατόφλι του 75%. Εάν όμω υπάρχει λιγότερη ε, φτώχεια, νομίζω πως μπορούμε εκεί πέρα να κάνουμε κάποια ε, εξοικονόμηση και τα λεφτά τα οποία εξοικονομούμε να πάνε π.χ. σε μια διασύνδεση των διαρθρωτικών ταμείων με τα διευρωπαϊκά δίκτυο. Αυτό το εξετάζει αυτή τη στιγμή η Επιτροπή Περιφερειακών ε, Θεμάτων καθώς επίσης και το θέμα αυτής της ενδιάμεσης κατηγορίας η οποία προτείνεται νομίζω πως η κυρία Κρέμπτ εδώ πέρα έχει φρούδες ελπίδες όσον αφορά τον συμβασμό στην Επιτροπή μας. Εγώ δεν θεωρώ πως θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η ενδιάμεση κατηγορία και δεν νομίζω πως χρειάζονται και ιδιαίτερη ενίσχυση ή πλουσιότερες περιοχές. Εδώ πέρα δηλαδή έχουμε πρόσκληση για σπατάλημα του χρήματος εγγυόμαστε μια μόνιμη επιδότηση για όλες τις ε, περιοχές. Κυρίες και κύριοι, αυτό το σύστημα δεν πρέπει να συνεχιστεί στο μέλλον. Γι' αυτό θα θέλαμε να διαγραφεί η παραγραφη 73, κατά τα λοιπά η έκθεση είναι μια χαρά. Υπάρχει μία μπλε κάρτα, γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Πίπερ κατά πόσο δέχεται μία ερώτηση από το συνάδελφό του. Δέχεστε μία ερώτηση από την κυρία Σουέτερ. Έχετε 30 δευτερόλεπτα για να υποβάλλετε την ερώτησή σας. Δεν λειτουργεί το μικρόφωνο σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ερώτημά μου απευθύνεται στον κύριο Πίπερ. Μιλάει για το ότι ονειρεύεται συνένεση η κυρία Κρέλ. Νομίζω πως υπήρχε μεγάλη πλειοψηφία στη ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιφερειακών Θεμάτων και νομίζω πως θα υπάρξει και στην Ολομέλη γιατί υπάρχει πλειοψηφία για την αλληλεγγύη μεταξύ των περιφερειών. Και θα ήθελα να μάθω γιατί περιέγραψε ως όνειρο αυτή την πλειοψηφία. Ευχαριστώ κύριε Πίπερ. Θέλετε να μας εξηγήσετε. Κοιτάξτε, αυτή είναι η δική σας ερμηνεία, κυρία Σρέντερ. Εμείς προτείναμε άλλο κείμενο στην Επιτροπή από αυτό το οποίο υπάρχει στην έκθεση τώρα Γκαρίγκα. Το πρώτο είναι αυτό. Και δεύτερον, εντός των πολιτικών σχηματισμών υπάρχουν ακόμα σοβαρές αντιρρήσεις επί της αρχής κατά της ενδιάμεσης κατηγορίας, το ξέρετε. Και πραγματικά είναι όνειρο το να λέει κανείς πως επιτύχαμε ε, συμβιβασμούς. Εξάλλου δεν ε, ξέρουμε ακόμα το τι θα γίνει στον Ομίλιο και απορώ με τη μεγάλη σας αισιοδοξία. Η κυρία Εστέλ Γκρελιέ έχει το λόγο. Η συζήτηση για τις δημοσιονομικές προοπτικές της Ένωσης το περιεχόμενό της, του στόχου της, περιγράφεται σωστά από αυτή την έκθεση της οποίας το κύριο προσόν είναι ότι καθορίζει ακριβώς στρατηγικούς στόχους και και για κάθε κράτος μέλος που μπορεί να έχει πιο περιορισμένες προσδοκίες. Ορισμένα κράτη-μέλη θέλουν να μειώσουν τη συμβολή τους, άλλα να την αυξήσουν και η έκθεση αυτή μιλάει ακριβώς για μια ολοκληρωμένη ενωσιακή πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη και το ιστορικό και τις νέες δικαιοδοσίες της Συνθήκης Λισαβόνας. Η έκθεση αυτή λοιπόν πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου πρέπει να αποτελέσει τη βάση της μελλοντική μας συζήτησης παρά το ότι είναι υπερβολικά ίσως φρόνιμη. Το 5% είναι όντως κάτι καλύτερο από αυτό που ζητούν ορισμένα κράτη-μέλη, αλλά το βασικό θέμα είναι πού θα μπει το όριο προς τα πάνω. Η πολιτική λιτότητα, η απογοήτευση των πολιτών είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και της κυκλικής κρίσης. Θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα τη σημασία που θα είχε η δημιουργία μιας ενδιάμεσης κατηγορίας περιφερειών για την κατανομή των περιφερειακών κονδυλίων πιο δίκαια. Καταλήγω λέγοντας ότι πρέπει να καταλήξουμε στη φορολόγηση της κερδοσκοπίας που θα ενδυναμώσει την εμπιστοσύνη στους πολίτες και θα βελτιώσει τα οικονομικά μας. Για δύο λεπτά ο συνάδελφος Χούκμαρκ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή γιατί τόνισε όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και επίσης χαίρομαι για το σαφές του συμπέρασμα που ζητάει σημαντικές αυξήσεις για την έρευνα και την επιστήμη γιατί είναι μία από τις προτεραιότητές μας αυτή. Θα ήθελα να δηλώσω και το δηλώνω προς την Κομισιόν ιδιαίτερα ότι η πολιτική ηγεσία είναι θέμα καθορισμού προτεραιοτήτων. Χωρίς προτεραιότητες δεν υπάρχει ηγετικός ρόλος, ούτε καθοδήγηση. Πάντοτε υπάρχουν ορισμένοι στόχοι σημαντικότεροι από άλλους. Αυτό ισχύει και για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και των χωρών μελών. Πρέπει οπωσδήποτε να αυξηθούν τα κονδύλια για την έρευνα, αλλά επίσης και για την επιστήμη γενικότερα. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας το θέμα της ανάπτυξης των αγροτικών αγορών, των αγορών των γεωργικών προϊόντων. Όμως κύριε Πρόεδρε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι προτεραιότητες είναι κάτι που πρέπει να καθοριστούν σε όλα τα επίπεδα, και στο ενωσιακό και στο εθνικό. Και εγώ δεν είμαι από αυτούς που επικρίνουν συστηματικά την Ένωση, αλλά ούτε και από εκείνους που επικρίνουν τα κράτη-μέλη, γιατί έτσι μειώνουν τη σημασία της δαπάνησης χρημάτων από εθνικές δικαιοδοσίες για συντάξεις, υγειονομική περίθαλψη. Εδώ δεν πρόκειται για αντίφαση μεταξύ κρατών μελών και ένωσης, αλλά για αγώνα κυριάρχησης και προτεραιοτήτων. Αν δεν καθορίσουμε σωστά τις προτεραιότητες μας δεν θα παίξουμε ηγετικό ρόλο και πρέπει να σας πω ότι αν δεν καταλαβαίνουμε τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα κράτη-μέλη, τότε δεν καταλαβαίνουμε την πραγματικότητα των πολιτών. Πρέπει να καθορίσουμε προτεραιότητες και όχι απλώς να αυξάνουμε προϋπολογισμούς. Γι' αυτό κύριε Επίτροπε, επιδείξτε πνεύμα ηγετικό, πάρτε πρωτοβουλίες, η έρευνα, οι υποδομές είναι από τις κύριες μας προτεραιότητες, διακόπτεται ο εισηγητής. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Κοτσολίνος. Αγαπητοί συνάδελφοι, ψηφίζουμε ένα στρατηγικό έγγραφο μεγάλης εμβέλειας που θα διέπει τις δημοσιονομικές προοπτικές μετά από το 2013. Μιλάμε για συνοχή μεταξύ στόχων και μέσων ως προς το νέο ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουμε και με βάση τη χρηματοοικονομική κρίση. Έτσι θα επενδύσουμε. Η συνοχή σημαίνει ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις ανάγκες καινοτομία που ζητά η κοινή γνώμη έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη και τις κοινωνικές παραγωγικές δυνάμεις. Το θέμα της συνοχής είναι ύψης της και ζωτικής σημασίας για να δούμε τι θα διαδραματίσει η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Η πείρα μας δείχνει ότι η συνοχή αποτελεί τον, την πεμπτουσία των σχεδίων μας. Θα πρέπει να δούμε τι θα, πού θα καινοτομήσουμε και πώς. Μιλάμε για την εισαγωγή μιας ενδιάμεσης κατηγορίας. Αυτό διότι σε πολλές περιπτώσεις τα χρόνια χρηματοοικονομικής κρίσης κατέδειξαν την ανάγκη μιας μεγαλύτερης υποστήριξης για τις περιφέρειες που δεν είναι τόσο αναπτυγμένες στην Ευρώπη, έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε την κατασπατάληση του χρήματος και να προωθήσουμε μια αναπτυξιακή πολιτική. Νομίζω με τη, με ρήτρα διασφάλισης ακριβώς αυτό επιτυγχάνουμε, δηλαδή εγγυόμαστε την επιβίωση των ενδιάμεσων κατηγοριών έτσι ώστε να υπάρχει πιο εξισορροπημένη ανάπτυξη την οποία θα πρέπει να εξασφαλίσουμε για την Ευρώπη για το μέλλον. Ο κύριος Έγγελ για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, τα 500 600 εκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν το 8% του παγκοσμίου πληθυσμού. Το 2050 θα είμαστε ε, ένα 5 με 6 παραπάνω και στη συνέχεια 3% επιπροσθέτως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσο μπορούμε να υποστηρίξουμε 2.000, 2.000 πρεσβείες, χιλιάδες στρατούς και ούτω καθεξός, καθεξής. Νομίζω ότι η Κίνα δαπανά πολύ χρήμα ακριβώς για να μπορέσει να υποστηρίξει να υποστηρίξει και να υποδεχθεί αυτές τις ε, δυσθεώρητα μεγάλες αντιπροσωπείες που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν ε, λάβετε υπόψη το 1,8% παραπάνω δια 30 αντιπροσωπείες, αυτό είναι παράλογο. Θα έχουμε μεγάλα χρέη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε να υποστηρίξουμε ένα 2,5% δηλαδή το 1,4% των εθνικών δαπανών. Ακόμα και όμως αυτό δεν επαληθευτεί, τι θα γίνει με τους ίδιους πόρους. Πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το 2,5% των δημοσίων δαπανών που θα πρέπει να υποστηρίξουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να θέσουμε σε εφαρμογή τη στρατηγική 2020 και για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το μεγάλο κληροδότημα της συνθήκης της Λισαβόνας. Δεν το έχουμε επινοήσει εμείς, το επινόησαν τα κράτη-μέλη. Με βάση αυτή την πραγματικότητα η έκθεση Γκαρίγκα είναι ε, μετριοπαθής αλλά είναι σχετικά φιλόδοξη σε σχέση με αυτούς που θέλουν να μας περιορίσουν ακόμα περισσότερο και γι' αυτό θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή την έκθεση. Ευχαριστούμε. Για 1,5 λεπτό. Ε, λεπτό έχει το λόγο ο κύριος Νταρντέν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτή η έκθεση είναι πολύ σημαντική για το μέλλον της Ευρώπης που θα πρέπει να είναι αλληλέγγυα και φιλόδοξη, ιδιαίτερα σε σχέση με τις ε, κρίσεις που αντιμετωπίσουμε. μέσα στα πλαίσια μίας, ενός νέου φιλελευθερισμού από πλευράς κρατών βλέπουμε ότι δεν επενδύουμε στις μεγάλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πάγωμα αυτό αυτού του προϋπολογισμού θα είναι επιζήμιο στην ανάπτυξη, σε αντίθετα από αυτό που πιστεύουν πολλοί. Ε, μια αύξηση του 5% θα πρέπει να είναι ένα ελάχιστο όρο έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε τη στρατηγική 2020, ιδιαίτερα με βάση τους κοινωνικούς στόχους και την καταπολέμηση των πλέον ενδεών. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή την αλληλεγγύη δημιουργώντας ενδιάμεσες περιφέρειες έτσι ώστε η πολιτική συνοχής να μπορέσει να καλύψει εδαφικά ολόκληρη την Ευρώπη. Ένα άλλο ε, παράδειγμα είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αντιμετώπισης της Παγκοσμιοποίησης που, ε, που μας απασχόλησε και απασχολεί και αυτή την έκθεση. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν αυτού του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε το πλαίσιο ως άχθος για τους εθνικούς προϋπολογισμούς αλλά ότι θα αποτελέσει προστιθέμενη αξία για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Το λόγο έχει η κυρία Γιαννάκου για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, η συνθήκη της Λισαβόνας δημιούργησε νέα πεδία αρμοδιότητας και ενίσχυσε τις πολιτικές της Ένωσης, γεγονός που αντανακλάται στη διαμόρφωση του επομένου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου της περίοδου 13-20. Συγχαίρω τον εισηγητή κύριο Γκαρίγκα για την ολοκληρωμένη έκθεσή του που απεικονίζει τις πολιτικές προτεραιότητες μιας ευρώπης διαφορετικής από αυτή που γνωρίζαμε με δεδομένες τις μεγάλες εσωτερικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ίδια η ένωση αλλά και οι πολίτες της και λαμβάνοντας υπόψη τον ενισχυμένο διεθνή της χαρακτήρα αντιλαμβανόμαστε ότι κύριος στόχος της πολιτικής πρέπει να είναι η μείωση των υφισταμένων κοινωνικών οικονομικών και εδαφικών ανισοτήτων. μια προβεβλημένη και επιτυχής πολιτική συνοχής αποτελεί από μόνη της ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και πρέπει να αποβαίνει προ όφελο όλων των κρατών μελών τη Ένωση. το νέο πρόγραμμα λοιπόν και το νέο πλαίσιο επταετού διάρκεια θεμελιώνεται στι δράσει τη στρατηγική 2020 είκοσι και έχει ως γνώμονα την ανάκαμψη τη Ευρώπη από την κρίση με την προώθηση έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. πολιτικές προτεραιότητε και στόχοι ορίζονται η προώθηση τη απασχόληση η ενίσχυση της καινοτομία η έρευνα η ανάπτυξη η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής η βελτίωση των επιπέδων εκπαίδευσης η κοινωνική ένταξη και η καταπολέμηση της φτώχειας. επίσης οι πολιτικές για τη μετανάστευση και εξασφάλιση πόρων για την ανάπτυξη δύσβατων και ακριτικών περιοχών. ο προϋπολογισμός της ένωσης αποτελεί τον κύριο μηχανισμό ενεργοποίησης της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών και ισχυρό εργαλείο μιας μεταρρύθμισης που θα μπορούσε να κινητοποιήσει πρόσθετους ιδιωτικούς και δημόσιους πόρους για να υποστηριχθούν οι επενδύσεις που θα λειτουργούσαν ως καταλύτης όσον αφορά την πολλαπλασιαστική επίδραση των δαπανών της ένωσης. ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να αυξηθεί κύριε πρόεδρε και να βασιστεί σε πραγματικούς ιδίους πόρους αν θέλουμε μια ευρώπη ισχυρή για τους πολίτες της και εναντί όλου του κόσμου ο προϋπολογισμός τη ένωσης είναι εργαλείο λοιπόν συνολικής και ολοκληρωμένης ανάπτυξης σε μια στιγμή που τα κράτη μέλη μόνα τους δεν μπορούν να για 1,5 λεπτό η κυρία Οκονή. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, συχνά λέμε ότι το χρήμα είναι η βάση του πολέμου, είναι όμως η βάση και της ειρήνης όπως του ευρωπαϊκού σχεδίου. Αν η Ευρώπη θέλει πραγματικά να εφαρμόσει τα προγράμματα που προβλέπει η συνθήκη ακόμη και, τα πιο και η πιο πρόσφατη μορφή της όπως της Λισαβόνας πρέπει να έχει τους απαραίτητους πόρους για να εφαρμόσει τους στόχους αυτούς. Επομένως είμαι υπέρ της αντίληψης των ιδίων πόρων και της δημιουργίας ενός φόρου για τις δοσοληψίες αυτή, μια τέτοια αύξηση του προπολογισμού θα πρέπει να συνοδεύεται από σημαντικέ εξοικονομήσει μέσω της βελτιστοποίηση των δαπανών. Παραδείγματο χάρη, μια πραγματική εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας, κοινή άμυνας, θα μπορούσε να διασφαλίσει μεγαλύτερη επιρροή της Ευρώπης διεθνώς, αλλά επίσης καλύτερη εκμετάλλευση των διαθεσίμων πόρων. Η έκθεση Γαρίδα Πολέδο είναι πολύ σημαντική σχεδόν ιδρυτικό σχέδιο της μελλοντικής ανάπτυξης της Ένωσης. Εκτός αυτού αναφέρει ότι δύο βάσεις μέχρι τώρα πολιτικής όπως η ΚΑΠ είναι κάτι που πρέπει να συνεχιστεί και δεύτερον η πολιτική συνοχής που είναι το κυριότερο χρηματοδοτικό μας εργαλείο για την επίδειξη της οικονομικής μας αλληλεγγύης. Πρέπει να ενδυναμωθούν όλα αυτά μέσω της δημιουργίας μιας ενδιάμεσης κατηγορίας περιφερειών ώστε να... Α, με συγχωρείτε κυρία Οκονή, τελείωσε ο χρόνος σας. Η κυρία Χιούμπνερ τώρα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, θα ήθελα να πω λίγα λόγια για την ανάγκη του να πάμε σε μια μεταρρύθμιση των ιδίων πόρων. Θεωρώ πως ο κυρίαρχος ρόλος ε, του ΑΕΠ ε, νομίζω κάνει λιγότερο αποτελεσματικό τον ε, κοινοτικό προϋπολογισμό, οδηγεί σε απαιτήσει να παγώσει και οδηγούμαστε στη λογική των διαπραγματεύσεων του 2011, ότι δηλαδή πρέπει να εφαρμοστούν όσα ίσχυσαν για τους εθνικούς προϋπολογισμούς και στον κοινοτικό. Αλλά δεν είναι ε, καθόλου προφανές πως ε, με ιδίους πόρους θα υπάρχει επανάσταση στην δυνατότητα χρηματοδότησης της Ένωσης. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν... Ε, αυτές τις αποφάσεις στο Συμβούλιο να τις ε, ψηφίσουν οι ίδιες χώρες και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει λοιπόν να πάμε πιο κοντά στις προσδοκίες των πολιτών. Αυτές οι επιτυχίες των εθνικών πολιτικών που επιστρέφουν από τις Βρυξέλλες δεν θα πρέπει να βασίζονται στο ότι πληρώνουν λιγότερα στο κοινοτικό προϋπολογισμό αλλά στο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραδείγματος χάρη θα χρηματοδοτήσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις για καινοτόμα έργα. Είναι σαφέ ότι θα πρέπει να υπάρχει επίση πλήρη διαφάνεια. Αυτό γίνεται εύκολο με έναν μόνο φόρο, αλλά μπορούμε να έχουμε και περισσότερου φόρους που θα ε, εκπληρώνουν τα κριτήρια τη ε, εναρμόνιση δικαιοσύνη, αποτελεσματικότητα κτλ. Η κυρία Καρβάλιο έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπο, θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον εισηγητή διότι έλαβε υπόψη τις βασικές προτεραιότητες που συνάδουν με την στρατηγική 2020. Μιλάμε για την ανάπτυξη που θα είναι επίκεντρο των ευρωπαϊκών πολιτικών. Χρειαζόμαστε καλύτερη και περισσότερη Ευρώπη. Γι' αυτό θα πρέπει να αξιολογήσουμε τους τομείς που βοηθούν στην ανταγωνιστικότητα όπως οι επιστήμες, η ενέργεια και η έρευνα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την έρευνα και ανάπτυξη καθώς και την ε, καινοτομία μέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής αριστείας. Επίσης θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε την έρευνα έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα 3% του ΑΕΠ που είναι ο απότερος στόχος. Επίσης θα πρέπει να υποστηρίξουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα, την υποστήριξη των υποδομών και ιδιαίτερα των υποδομών ενέργειας, έτσι ώστε να ε, έχουμε τους κατάλληλους όρους για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ για να βοηθήσουμε για τον ηγετικό χαρακτήρα της Ευρώπης ανά τον κόσμο. Ευχαριστούμε την κυρία Καρβάλιο. Η κυρία Μπάρμπαρα Ματέρα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή για την εξαιρετική του εργασία που τον απασχόλησε εδώ και ένα χρόνο και, έφτασε, και όπου έφτασε σε μεγάλη συνένεση. Φτάσαμε όχι σε επίλυση της κρίσης αλλά ε, διατρανώσαμε το ρόλο μας μέσα στα πλαίσια της παγκόσμιας κακέρας. Επίσης η έκθεση αυτή συνάδει με τη στραγητή 2020 καθώς και με τα προαπαιτούμενα της συνθήκης της Λισαβόνας. Χρειάζεται λοιπόν η δημοσιονομική προσαρμογή. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ενέργεια, τις μεταφορές, την έρευνα και ανάπτυξη, την κατάρτιση, τις πολιτικές υπέρ των νέων, θα πρέπει όλες αυτές οι πολιτικές να ενταχθούν στους μελλοντικούς μας προϋπολογισμούς, ενώ οι βασικοί πυλώνες της συνοχής και της ΚΑΠ θα πρέπει να ε, αρκεστούν στο παρόν επίπεδο χρηματοδότησης. Η Ευρώπη με τους μεγάλους στόχους ε, λαμβάνει υπόψη τους ποσοτικούς περιορισμούς από εθνικής πλευράς, γι' αυτό θα πρέπει να συμμετάσχει και ο ιδιωτικός τομέας μέσα ε, μέσα στα πλαίσια της ε, συνέργειας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Βλέπουμε με ανησυχία τις ε, προτάσεις ε, εισδοχής των ενδιάμεσων περιφερειών, όπως ζητάει και η Ιταλική κυβέρνηση, που θα πλήξει τις περιφέρειες αυτές. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει πλήρης χρηματοδότηση με βάση τους ίδιους πόρους και είναι ο μόνος τρόπος για να εγγυηθούμε το μέλλον και την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Η κυρία Τσίκαου νομίζω ότι έχει σηκώσει μια, την μπλε κάρτα. Θέλει να υποβάλει μια ερώτηση ή θέλετε να εγγραφείτε για το Catch the Eye, κυρία Τσίκαου. Δεν σας ακούω κυρία Τσικάου. Για το catch the εντάξει. Η κυρία Γκρέσλε για ένα μισή λεπτό. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συναδελφοί, μαζί με το πακέτο των πολιετών δημοσιονομικών προοπτικών έχουμε και το καθεστώς του προσωπικού. Αυτά αναφέρονται στις παραγράφους 25 ε, και 126. Σας παρακαλώ να τα κοιτάξετε πάρα πολύ έντονα αυτά κύριε Επίτροπε γιατί το τι κάνουμε έχει εξίσου μεγάλη σημασία με το πώς το κάνουμε και θα πρέπει να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή όλων αυτών των προγραμμάτων του προγράμματος 2020 κτλ. Θέλω η Κομισιόν να προβλέψει ισχυρότερο ρόλο για τον εαυτό της και να μην δώσει όλες τις λειτουργίες της σε εξωτερικούς. Οπότε θα πρέπει να προβλέψετε νέες θέσεις για τις νέες αποστολές που ε, η Κομισιόν ε, θα επομιστεί. Επίσης, ε, ξέρετε πως έχουν μέχρι και πάρα πολλές αργίες, μέχρι και 13 ημέρες αργίας οι οποίες προβλέπονται. Πρέπει λοιπόν να τις μειώσετε αυτές για να ε, μπορέσουμε να έχουμε αποτελεσματικότερη λειτουργία της διοίκησης για την Ευρώπη 2020. Αυτό νομίζω πρέπει να το κάνει και ο πρόεδρος της Κομισιόν και η Κομισιόν στο σύνολό της. Ευχαριστώ για 1,5 λεπτό. Κυρία Κεντρεζιεύσα. Ποσδάνια βιολολέτνιχ ραμ φινανσόβιχ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι πρόκειται για μια εξαίρετη έκθεση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, μια έκθεση την οποία είχαμε υποστηρίξει στην Επιτροπή σου. Ελπίζω λοιπόν η έκθεση αυτή να αποτελέσει μια σημαντική βάση για τις ε, διαπραγματεύσεις για το μελλοντικό πολιετές ε, μουσιονομικό πλαίσιο και χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν να στηρίξουν την ε, τροπολογία μου για την πολιτική υπέρ των νέων σε καιρό που οι νέοι Ευρωπαίοι είναι ένα από τα βασικά θύματα της οικονομικής κρίσης θα πρέπει να υποστηρίξουμε πρωτοβουλίες που στόχο έχουν να βελτιώσουν την ε, πρόσβασή τους στην ε, εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας. Γι' αυτό προγράμματα όπως νέοι σε δράση και διαβίου κατάρτισης έχουν χαμηλό κόστος ανασυμμετέχοντα και είναι πολύ αποτελεσματικά και πρέπει να αποτελέσουν ε, στοιχείο και των μελλοντικών δημοσιονομικών προοπτικών και βεβαίως να έχουν περισσότερη χρηματοδότηση. Ταυτόχρονα θα ήθελα να πω πως είμαι ικανοποιημένη για το ότι έχει διατηρηθεί η χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής γιατί είναι μια πολιτική η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για την εφαρμογή της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020 αλλά στόχο έχει να εμβαθύνει την ολοκλήρωση και την αλληλεγγύη στην Ευρώπη με το να μειώσει τις υπάρχουσες διαφορές στην Ευρώπη. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Τελειώσαμε με τον κατάλογο εγγεγραμμένων ομιλητών και τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία Catch the Eye. Έχουμε 19 συναδέλφους εγγεγραμμένους. Θα δώσω το λόγο 8, σε 8. Δεν μπορούμε να τους υπερβούμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να ακούσουμε και τον εισηγήτη και τον ε, ε, Επίτροπο πριν μπουν 700 συνάδελφοι για να ψηφίσουν. Θα σας διακόψω ακριβώς πάνω στο λεπτό να το ξέρετε αυτό. Καταρχήν, έχει το λόγο ο κύριος Νικουλέσκου. Ε, ευχαριστώ. Ο εισηγητής μίλησε για την ανάγκη να μπορέσουμε να διασυνδέσουμε τις ανάγκες μας με τις προτεραιότητές μας. Διαφορετικά ε, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτά τα πλαίσια. Θα ήθελα να δεχτώ το όραμα που διέπει την ΚΑΠ και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ορισμένες βασικές ιδέες. Να κρατήσουμε την ΚΑΠ στα ίδια επίπεδα για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο και να λάβουμε υπόψη τον ρόλο της γεωργίας. Χρειάζεται να προσαρμόσουμε και τον προϋπολογισμό. Επίσης θα πρέπει να κρατήσουμε την ε, ΚΑΠ στα ίδια πλαίσια έτσι ώστε να προωθήσουμε τις αγροτικές περιοχές μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής 2020. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και μία αναθεωρημένη ΚΑΠ έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε πιο αποδυτικά τον προϋπολογισμό για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις νέες ανάγκες που δημιουργούνται. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Μπαλτσίτη. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους του ηγητέ για τη δουλειά που έκανα. Σήμερα έχουμε μια σαφή θέση του Κοινοβουλίου για τις προσδοκίες των πολιτών και για τις δημοσιονομικές πρόπτικες. Θα πρέπει να αλλάξουμε την πολιτική μας και την κατεύθυνσή μας και αυτό φαίνεται στη στρατηγική 2020. Πρέπει να υπάρχει μια ενιαία αγορά ενέργειας, να δεσυνδεθεί η Ευρώπη από πλευράς μεταφορών και να μειωθούν οι ανισότητες μεταξύ των περιοχών της ε, Ένωσης. Επίσης χρειάζεται σωστή γεωργική πολιτική. Υπάρχουν και άλλοι τομείς οι οποίοι είναι αναγκαίοι για να δημιουργήσουμε ανταγωνιστική Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης τεράστιες επενδύσεις στην εκπαίδευση. Πρέπει λοιπόν να βρούμε νέες πηγές χρηματοδότησης και ο φόρος ε, αυτός στις ε, χρηματοοικονομικές αναλλαγές είναι μια τέτοια δυνατότητα. Ευχαριστώ κύριος Γιάννη Euh, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ένα από τα θέματα τα οποία προέκυψε στη συζήτηση είναι ποια ακριβώς είναι η ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Ελπίζω λοιπόν πως η Κομισιόν θα μπορέσει να εξηγήσει γιατί τα διάφορα σημεία του προπολογισμού έχουν κάποια ιδιαίτερη προσθέμενη αξία. Και αυτό νομίζω ε, είναι σωστό για να ξέρουμε και γιατί ακριβώς ε, ψηφίζουμε δεύτερον. Υπάρχει και η συζήτηση των ιδίων πόρων. Ε, έχουμε και την απόφαση του 1984 για την Βρετανική επιστροφή είναι δυνατόν να διαρκέσει επάπειρον. Είτε δεν θα υπάρχει επιστροφή για κανέναν, είτε χώρες οι οποίες θα είναι στην κατάσταση που ήταν η Βρετανία το 1984 να έχουν την ίδια μεταχείριση. Αυτά και σας ευχαριστώ. Μάλιστα. En primer lugar, más Europa γιατί ψάχνουμε πάντα να βρούμε να αυξήσουμε πόρους εμείς θέλουμε καλύτερη Ευρώπη και ορισμένοι θεωρούν ότι αυτό σημαίνει λιγότερες δικαιοδοσίες για τα κράτη-μέλη. Ένας προπολογισμό όμως πρέπει να λαμβάνει υπόψη του όλες τις πτυχές των οικονομικών θεμάτων. Παραδείγματος χάρη υπάρχουν στρατιωτικές δαπάνες και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Ο κύριος Λεβαντόφσκι βλέπω ότι χαμογελάει. Αυτό είναι λυπηρό λόγω της κατάστασης που αντιμετωπίζουμε. Πώς γίνεται, πώς γίνεται λέγω, πώς γίνεται να θεωρήσουμε σωστό να πληρώνουν οι πολίτες για την κρίση ενώ ταυτόχρονα μειώνονται οι κοινωνικές δαπάνες κλπ. Επόμενος Ρούμπιχ. Ευχαριστώ. Εξακολουθεί να μην δουλεύει το μικρόφωνο μου, γι' αυτό άλλαξα θέση και σβήνει το μικρόφωνο του μιλητή. Ο κύριος Ρούμπιξ έχει το λόγο. Ρούμπιξ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους ε, συναδέλφους μας το εξής. Όταν μιλάμε για τον προπολογισμό πρέπει να θυμόμαστε πως ε, οι Ευρωπαίοι πολίτες γίνονται όλο και πιο επιφυλακτικοί ε, απέναντί μας. Οπότε δεν πιστεύω πως ο προϋπολογισμός είναι εναρμονισμένος με τους φιλόδοξους στόχους ε, που υπάρχουν στρατηγική του 2020. Ένα άλλο ερώτημα. Εσείς ε, κύριε Επίτροπε υποσχεθήκατε στους λετονούς αγρότες να εναρμονίσετε τις άμεσες ενισχύσεις ε, βεβαίως αν εγκριθεί ο προϋπολογισμός αυτός δεν μπορείτε να εκπληρώσετε αυτή την υπόσχεσή σας. Θα ήθελα λοιπόν μια φορά να λάβουμε υπόψη και τα συμφέροντα των ψηφοφόρων μας. Ε, Andrew Bronze. Ευχαριστώ κύριος Andrew Bronze. Ευχαριστώ. Μα νόμιζα ότι δεν μπορεί να γίνει χειρότερη η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι που διάβασα αυτή την έκθεση. Ξεκινάει έτσι με αρκετές ε, ψευδεστήσεις. Λέει ποτέ δεν ζητούσαν περισσότερα οι Ευρωπαίοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω, οι Βρετανοί ζητάνε να σηκωθούμε να φύγουμε, ίσως αυτό εννοεί. Επίσης, Έχουμε αύξηση του προπολογισμού μέχρι το 2013 και λέει πως ε, ακόμα και η αύξηση κατά 5% ε, λίγο θα συνεισφέρει στους στόχους Ένωσης. Ε, κάτι είναι και αυτό. Η παράγραφος 166 ζητάει να σταματήσουν οι επιστροφές ε, και βεβαίως αυτός είναι ο μηχανισμός με τον οποίο πληρώνουμε απλώς μια απαράδεκτη αντί για μια τελείως παράλογη ε, καθαρή εισφορά το Ηνωμένο Βασίλειο. Η 169 λέει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μπορεί να επιβάλλει φόρους χωρίς τη συνένεση και τον έλεγχό μας η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σικέρσκη. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι καταφέραμε να φτάσουμε σε έναν πολύ καλό συμβιβασμό γιατί η έκθεση αυτή αποτελεί μια συνέχεια και προτείνει και αλλαγές. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές θα πρέπει να είναι σταθερές έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε τον ίδιο προϋπολογισμό για τη συνοχή και την ΚΑΠ. Θα πρέπει επίσης να άρουμε τις διαφορές και αυτό θα μπορέσει να ευεργετήσει όλα τα κράτη-μέλη. Η ΚΑΠ ευεργετεί σε τελευταία ανάλυση όλους τους καταναλωτές. Οι αγρότες έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα, μην το ξεχνάμε αυτό, παρά τις, τη νέα υποστήριξη. Άρα θα πρέπει να υποστηρίξουμε την ε, κατάσταση της ΚΑΠ. Θα πρέπει να λάβουμε και την κατάσταση των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ. Ποιος θα καταβάλει το αντίτιμο. Ε, πο, δυστυχώς διακόπη ο μιλητής. Ο κύριος Σταυρακάκης έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Το Κοινοβούλιο στέλνει σήμερα ένα ξεκάθαρο μήνυμα τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και στους Πρωθυπουργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα προπολογισμό μέχρι το 2020 αντάξιο των ευθυνών τη αλλά και των προσδοκιών των πολιτών. Όσον αφορά την πολιτική συνοχή, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Ναι, σε μια πολιτική συνοχή με επαρκή χρηματοδότηση για να συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη, σε νέε θέσει εργασία, στην κοινοτομία ναι σε μια αυτόνομη πολιτική συνοχή ναι στο συντονισμό σε όλα τα επίπεδα χάραξη πολιτική από το στρατηγικό σχεδιασμό στην υλοποίηση ναι στη δημιουργία ενδιάμεση κατηγορία στήριξη περιφερειών ναι σε ειδικά μέτρα για νησιώτικε και ορεινέ περιοχέ τη ευρώπη αλλά επίση και δύο ξεκάθαρα σημαντικά όχι όχι σε οποιαδήποτε διάσπαση τη πολιτική αυτή σε διάφορου τομεί και τέλο όχι στην επιβολή κυρώσεων συνδεδεμένων με το σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη. Ευχαριστούμε. Λίγοι λοιπόν ο γύρος του Catch the Eye και ζητώ συγγνώμη στους 11 ή 12 συναδέλφους που είχαν εγγραφεί, όμως δεν υπάρχει χρόνος για τις παρεμβάσεις τους. Μπαίνουμε στην τελική φάση της συζήτησης, ε, δίνοντας το λόγο στον Επίτροπο, τον κύριο Λεβαντόφσκι, για να αντιδράσει στις 49 παρεμβάσεις των Ευρωβουλευτών. Κύριε Λεβαντόφσκι, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, έχω καταναλώσει όλο μου το χρόνο ήδη, αλλά γι' αυτό θα περιοριστώ σε δύο σύντομα σχόλια. Στην σημερινή διεθνή συγκυρία, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για την κακή διαχείριση εθνικών προϋπολογισμών, αλλά μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στις επενδύσεις ενώ οι εθνικοί προϋπολογισμοί αφορούν κυρίως θέματα κοινωνικής μεταφοράς πόρων. Αυτό που θα ήταν ρεαλιστικό θα ήταν μία προοδευτική μεταφορά. Και τέλος, προβλέπω εξ ονόματος της Κομισιόν η ψηφοφορία να ανταποκρίνεται στην ευρεία συνένεση που ακούστηκε εδώ στην αίθουσα ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αυξήσει την επιρροή του. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Λεβαντόφσκι. Τελειώνουμε με τον εισηγητή, τον κύριο Γαρίγα και Πολέδο για δύο λεπτά τον οποίο ούτως ή άλλως συγχαίρω εκ των προτέρων για την εργασία του. Δύο λεπτά λοιπόν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις εθνικές αντιπροσωπείες που αντιστάθηκαν, αντιστάθηκαν ως προς τις πιέσεις των κρατών μελών και θα υπερψηφίσουν αυτή την έκθεση. Νομίζω ότι δεν πρόκειται για μια συζήτηση για τον προϋπολογισμό κάθε αυτό, αλλά για την υπεροχή του κοινοτικού συστήματος και νομίζω ότι δεν τα κατάφεραν εκείνοι που θέλησαν να μειώσουν τον προϋπολογισμό, διότι θέλουν νέες προτεραιότητες και λιγότερο προϋπολογισμό. Έτσι θα καταφέρουν και λιγότερες προτεραιότητες και χαμηλότερο προϋπολογισμό. Άρα δεν νομίζω ότι μπορείτε να μιλάτε για μία διακυβερνητική προσέγγιση. Αφήστε το αυτό στο Συμβούλιο. Εσείς πρέπει να προασπιστείτε μία Ευρωπαϊκή Ένωση με τις προτεραιότητες και τις ευθύνες της και με έναν επαρκή προϋπολογισμό. Εμείς δεν θέλουμε να αυξήσουμε κατά ένα 5% τις ε, κοινοτικές δαπάνες. Θέλουμε ε, να ελαφρύνουμε τους εθνικούς προϋπολογισμούς και να λάβουμε υπόψη ορισμένες ε, υπερεθνικές δαπάνες οι οποίες μπορούν να καλυφθούν και να εκτελεστούν καλύτερα. Αυτή είναι η προστιθέμενη αξία της Ευρώπης που δέχτηκαν όλες οι ομάδες αυτού του σώματος στην Επιτροπή ΣΥΡ. Νομίζω ότι πρόκειται για μια πρόταση μεγάλης εμβέλειας, φιλόδοξη, που προαπαιτεί μεγάλη ε, ένα μεγάλο όραμα από τα κράτη-μέλη και αυτή είναι και η πρόκληση. Εδώ έγκυται η πρόκληση. Γι' αυτό ε, δέχομαι αυτές, ε, αυτή τη συζήτηση, τη ζωηρή συζήτηση, δείχνει το μεγάλο αυτό ψηφιδωτό εθνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και νομίζω ότι έχουμε εμπλουτιστεί, είμαστε πολύ πιο εμπλουτισμένοι από αυτή τη συζήτηση ως σώμα. Ευχαριστούμε. Κλείνει λοιπόν η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει μέσα σε λίγα λεπτά. Ευτυχώς τελειώσαμε με αυτή τη συζήτηση μίζωνος σημασίας και θα διακόψουμε για 3-4 λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι για την κατανόησή σας. Διακόπτουμε για τρία-τέσσερα λεπτα σας ευχαριστω πολυ κυριες και κυριοι για την κατανοηση σας διακοπτουμε για τρία λεπτα